Άουκεν. Μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών. Κυρία Σιγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μέρα για μας ε, που αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόταση γιατί μιλάμε για μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον με εκατοντάδες, εκατομμύρια λεπτές σακούλες που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο που καταλήγουν κατευθείαν στη φύση ως απορρίμματα και κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε το μέγεθος του προβλήματος. Βλάβες λοιπόν στην θάλασσα, στη φύση, στα πτηνά, σε όλα τα ζωά και θα πρέπει λοιπόν κάπως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Μιλάμε για ένα, το πρώτο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόληψη φυσικά είναι στην κορυφή. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται δράση. Εδώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρχικά δεν ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που είχαμε τώρα. Ήταν μάλλον ασθενής. Είχαμε διάφορους ευσεβείς πόθους και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την εξαιρετική συνεργασία. Καταρχάς τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν μαζί μου από την αρχή και για όλο τον δρόμο που ακολουθήσαμε. Τον κύριο Χερμπράνδη, τον συνάδελφο Λαβία, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί καταφέραμε να πετύχουμε μια πολύ καλή πρόταση που πέρασε. Και επίσης την Ιταλική Προεδρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και να τη συγχαρώ για την εξαιρετική προσπάθεια γιατί τώρα έχουμε μια κοινή θέση ενώπιον μας η οποία σημαίνει μία μείωση σημαντική. Το 2018 οι χώρες θα πρέπει να, έχουν, να θέσουν μία τιμή σε όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς και μετά το 2018 ελπίζουμε να έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο. Στην Ιρλανδία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος γιατί επισημάνθηκε η τιμή αυτής της πλαστικές τσάντες και έτσι υπήρξε μείωση 5%. Το... Ο στόχος λοιπόν είναι οι 90 λεπτές πλαστικές σακούλες ανά άτομο μέχρι το 2019 και 40 σε σακούλες μέχρι το 2025. Θεωρώ ότι είναι καλό αποτέλεσμα. Έχω εδώ ένα καλό φίλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δυστυχώς πρέπει να πω ότι εξ αρχής ήταν κατά ημών. Είχαν διάφορες ενστάσεις άσχετες, τις οποίες και προέβαλαν, για να μην κάνουν τελικά τίποτα. Έλεγαν ότι θα πρέπει οι χώρες να το κάνουν αυτό, αλλά δεν το κάνουν οι χώρες μόνος τους. Παρά λοιπόν τα μεγάλα οικονομικά παιχνίδια 740 ε, εκατομμύρια ευρώ ανά έτος ε, σύμφωνα με τις υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξοικονομηθούν. Παρά όλα αυτά, παρά όλα αυτά, είχαμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ξεχάσω το πρόσωπο του κ. Τίμερμαντς. Όταν ε, ελήφθη η απόφαση να μην αποσυρθεί η πρόταση, Τα τέσσερα λεπτά που πήρα το λόγο, χιλιάδες, ε, εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες τέτοιες πλαστικές ε, σακούλες καταναλώνονται στην Ευρώπη. 15.000. Να ευχαριστήσω όλες τις καλές δυνάμεις εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνέβαλαν και πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ότι κάτι κάνουμε γιατί είναι πραγματικά μια αμοιβαία εποφελής κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ η κυρία Άουκερ, κυρία, κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλημέρα. Σήμερα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την τελευταία φάση της νομοθετικής διαδικασίας, να αθετήσουμε δηλαδή μια οδηγία που έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση σειρά σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η υπερβολική κατανάλωση και η μόλυνση μέσω των πλαστικών σακουλών. Αυτές οι σακούλες όπως αναφέρθηκε πολύ εύκολα ξεφεύγουν από τη διαχείριση των αποβλήτων και συσσωρεύονται στο περιβάλλον και πολύ συχνά υπό τη μορφή και θαλασσίων αποβλήτων. Από τη στιγμή που αποβάλλονται μπορεί να διατηρηθούν εκατοντάδες χρόνια ακόμα και σαν μικροσκοπικά μόρια που απειλούν το περιβάλλον σε όλο τον κόσμο, κυρίως το θαλάσσιο περιβάλλον, σαν θαλάσσια απόβλητα. Αυξάνεται η κατανόλωση των πλαστικών σακουλών περίπου 100 δις σακούλες το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι 200 σακούλες κατά άτομο το έτος. Αυτό συνεπάγεται και σπατάλη πόρων και έχουν γίνει σύμβολο μιας κοινωνίας των σκουπιδιών και σύμβολο μη βιώσιμου τρόπου ζωής. Οι ελαφρές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που χρησιμοποιούνται άπαξ και μετά πετιόνται είναι ένα παράδειγμα ενός γραμμικού μοντέλου αντιμετωπίσεως των πόρων μας. Χρειάζεται λοιπόν κάτι να γίνει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της θαλάσσιας ρήπανσης. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε πλαστικά απόβλητα αυτή η ρήπανση και πρέπει να διασώσουμε τους πόρους και να έχουμε ανακυκλούμενη κυκλική οικονομία δηλαδή. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται δράση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό όμως να κάνουμε αυτό που μας ανήκει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση για τη συσκευασία και την οδηγία για τα απόβλητα συσκευασία και για να μειώσουμε την ε, χρήση των πλαστικών σακουλών μπορεί να επισημοποιηθεί σήμερα. Βλέποντας τις διάφορες θέσεις των συνομοθετών στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας βλέπουμε σαφώς ότι δεν ήταν εύκολη δουλειά αλλά χάρη στις προσπάθειες που ανελήφθησαν από όλα τα μέρη τώρα έχουμε ένα συμβιβασμό μπροστά μας Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την εισηγήτρια την κυρία Μαργαρίτα Όκεν για τη δουλειά που έκανε βάσει της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τους κοιόδης εισηγητές της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη συμφωνία που πετέχθη από τους συνομοθέτες παρόλο που συμπεριλαμβάνει κάποια στοιχεία που κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν καλό να καλυφθούν ε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε διαφορετικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά αυτή η συμφωνία κατέστη εφικτή διότι έχουμε κοινό στόχο, δηλαδή περιορισμό της καταναλώσεως και της ρήπανσης από τις πλαστικές σακούλες. Το κείμενο που σας υπευλήθη σήμερα θα κάνει πραγματικά τη διαφορά όσον αφορά την επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Άουκεν. Νομίζω ότι κάναμε ένα σημαντικό ε, βήμα και έτσι θα απαλλαγούμε από κάποιες κακές καταναλωτικές συνήθειες. Το ανέφερε και ο κύριος Επίτροπος. 90% των πλαστικών σακούλων πετιούνται. Μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια τέτοιες ε, σακούλες οι οποίες καταήγουν στις χωματερές ή στη φύση γενικώ. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Την ευθύνη την έχουμε εμείς. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συνήθεια. Επομένως, θα πρέπει τώρα να ενεργήσουμε με τρόπο φιλικό προς τον πολίτη. Περί αυτού πρόκειται σήμερα. Όπως είπε η συγκέντρια, σε πολλές χώρες έχει βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί κανείς να διαλέξει. Ας πούμε, στην Ουγγαρία, ξέρετε, από το 2011 υπάρχει μια χρέωση για αυτές τις σακούλες και αυτό οδήγησε σε μείωση της χρήσης τους. Όλοι επομένως θα πρέπει κάτι να κάνουν. Μιλάμε για μέγεθος ε, που φτάνει στα 15 μικρά. Άρα θα πρέπει να δούμε που θα καταλήξουμε πάνω σε αυτό να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό και να βρούμε τελικά έναν τρόπο να έχουμε ένα πιο ε, υγιές περιβάλλον. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να λάβουμε κάποια απόφαση. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Χόλβενη, από τον κύριο έχετε ε, Μπλε κάρτα. Αποδέχεστε. Λαθέπτα. Αποδέχεστε. Έχετε το λόγο κύριε. Εδώ, εδώ είμαι. Εδώ, εδώ είμαι λέω ο υπερωτών. Αποδέχεστε την μπλε κάρτα μου κύριε Χόλβενη. Κύριε Χόλβενη. Very um, Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χολβενή, μας λέτε εδώ για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε και μας λέτε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε συμβασμό. Δεν νομίζω ότι για ένα θέμα ζωής και θανάτου θα πρέπει να συμβαστούμε. Είναι πάρα πολύ ρηπαντικό αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να ζητήσουμε από Συμβούλιο και Επιτροπή να απαγορεύσει, όχι να περιορίσει τη χρήση αυτών των σακουλών. Δεν συμφωνείτε. Χόλβενη. Σας ευχαριστώ που μου την ευκαιρία να διατυπώσω το ότι συμφωνώ 100% μαζί σας όμως εν προκειμένου νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα ο καθένας να καταβάλει μια προσπάθεια μέσα στη χώρα του και βεβαίως η Ευρώπη δεν πρέπει να τα κάνει όλα ε, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε τι έγινε μέχρι σήμερα. Εάν επομένως κάθε χώρα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που έχει και προχωρήσει γρηγορότερα και πιο μακριά, τότε θα τα ακολουθήσουν και άλλοι. Ο Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τη συγγήτρια την κυρία Άουκεν για την αποφασιστική δουλειά που έκανε στου τους μήνες. Αυτό που έχουμε τώρα μετά τις διαπραγματεύσεις που κράτησαν πολύ και που μπλοκαρίστηκαν επί της Ιταλικής Προεδρίας είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που ξεπερνά το συγκεκριμένο θέμα που υπενθυμίζαμε να υποχρεώσουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να μειώσουν τη χρήση των πλαστικών σακουλών που θεωρούνται ένας από τους παράγοντε ρήπανσης εν γέννη και πρώτος ε, τον παράγων για την θαλάσσια ρήπανση. Αλλά είναι συμβολική πτυχή κατά την άποψή μου αυτή η συμφωνία. Γιατί αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τα απόβλητα είχε ε, ήταν στη βάση σωστής διαχείρισης βιώσιμης το πρώτο R το ήταν το reduction δηλαδή μείωση της, ε, των αποβλήτων δεν λειτουργήσε Δώσαμε, είδαμε στην Ευρώπη ότι βλέπουμε ότι τα απόβλητα έχουν αυξηθεί αυτά τα χρόνια και τα χρόνια της κρίσης λόγω και έλλειψης να εφαρμόσουμε σοβαρές πολιτικές πρόληψης. Αυτό το κείμενο ξεκινά από εκεί. Δηλαδή για πρώτη φορά προσπαθούμε να κινηθούμε στο πρώτο επίπεδο των αποβλήτων. Να πούμε στα κράτη-μέλη θα πρέπει να μειώσουν την παραγωγή των αποβλήτων με στόχους υποχρεωτικούς με την εισαγωγή ε, μιας τιμής και περνά στο άλλο θέμα που κάνει τη διαφορά στο κείμενο. Με την οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο ώστε να προωθήσουμε την ανακυκλούμενη κοινωνία που είναι νέο σύνολο της βιώσιμης οικονομίας. Θέλουμε να μειώσουμε τα απόβλητα, σε αυτή την περίπτωση τις πλαστικές σακούλες και αυτό σίγουρα θα προωθήσει πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων με θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την όλη οικονομία. Περνάμε λοιπόν από προϊόντα μιας χρήσεως από τη γραμμική οικονομία προ μια λύση εναλλακτική που έχει λιγότερο αντίκτυπο και για τους πόρου και για το περιβάλλον και που τονώνουν και νέε τεχνολογίες πράσινες. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της πράσινης χημία για την παραγωγή των οργανικών σακουλών και θα ήθελα να κλείσω και να πω ότι είναι σημαντική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει και θα το κάνουμε ταχύτερα με νέα πρόταση πιο φιλόδοξη που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον όλον κύκλο των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καλώς ορίσατε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ορίσατε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν παρουσιάστηκε, γιατί θεωρώ ότι το θέμα των ε, πλαστικών σακουλών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ήταν αρκετά ευέλικτη αρχικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έδινε διάφορες ε, ε, εναλλακτικέ λύσεις στα κράτη-μέλη. Τώρα όμως το αποτέλεσμα είναι υπερβολικά δεσμευτικό. Το την επισήμανση, για παράδειγμα, για τις δύο αποκοδομήσιμες ε, σακούλες, δεν μπορώ να το αποδεχτώ, γιατί είναι μεγάλο το γραφειοκρατικό άχθος και για τα κρατημέλη και για τους ε, φορείς. Υπάρχουν διάφορα θέματα όπως ε, οι εκθέσεις για τις όξο πλαστικές σακούλες που με ανησυχούν. Ανησυχώ γιατί διάφορα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι προβληματικά όπως το θέμα της μη διακριτικής ε, και μη αναλογικής αντιμετώπισης καθώς και θέματα της λειτουργίας της ενέας εργα... Ε, αγοράς. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προορίζονται από την οδηγία, αλλά δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ε, και να τεκμηριώνουν τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Η κυρία Άουκεν, τέλο είπε ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε γιατί οι χώρες δεν κάνουν τίποτα από μόνε τους. Αυτό πολύ απλά είναι ψέμα γιατί στη δική μου χώρα ήμασταν κατά της έλλειψης ευελιξίας αλλά παράλληλα προτείναμε μέτρα για τη μείωση της πλαστικής σακούλας τα οποία πλέον έχουν περάσει. Άρα δεν ισχύει ότι άμα το κάνει η Ευρώπη δεν θα το κάνουν τα κρατη Το κάνουν και μάλιστα με το δικό τους ρυθμό, το οποίο αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χερμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμα και στα πιο απόμακρα μέρη του πλανήτη αυτού δεν βρίσκουμε πτηνά χωρίς πλαστικά στα στομάχια τους. Πλαστικά τα οποία δεν έχουν ε, δεν, έχει δεν έχουν χωνευτεί και συχνά είναι τοξικά και ξέρουμε αποτελούν ένα από το βασικό λόγο ρήπανσης με πλαστικό ή πλαστικές σακούλες και πολλά από αυτά τα θαλάσσια ζώα, τα πτήνα έχουν στα στομάχια τους κάποια από τις εκατοντάδες εκατομμύρια σακούλε που καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Παρά τα πολύ ανησυχητικά αυτά όμω θέματα υπάρχουν καλέ ειδήσει, δύο καλέ ειδήσει. Αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα καταρχά είναι εύκολο στην επίλυσή του. Παρά το γεγονό ότι είναι τεράστιο. Και κατά δεύτερον υπάρχει τεράστια υποστήριξη από το κοινό για να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό. Ω εκ τούτου το αποτέλεσμα το οποίο συζητάμε σήμερα αποτελεί θεωρώ ένα παράδειγμα πολύ καλής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είδαμε μια ένα ενωμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στην καλή εισηγήτρια την κυρία Άουκεν την οποία και ευχαριστώ. Αλλά επειδή επίσης είχαμε μια προεδρία, την Ιταλική, η οποία δεν εστιάστηκε απλά στο να αποφύγει τα προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά που πραγματικά ήθελε να επιλύσει ένα πρόβλημα. Κάτι το οποίο δυστυχώς είναι πρωτόγνωρο από πλευρά του Συμβουλίου. Αντίθετα με αυτά που ενδεχομένως πιστεύουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι εσείς κυρία Βέλα, αυτή η νομοθεσία στο μέλλον θα θεωρηθεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τελευταίων χρόνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Φορέντσα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω να σας πω ότι παρά αυτές τις απαραδεκτές πιέσεις από τα λόμπι των παραγωγών και διανομέων και παρά την αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ακριβώς ε, είπε και η συγκεντρία φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία ούτως ώστε τα μέσα χρόνια θα μειωθεί η χρήση και η κατανάλωση των τελαφρών σακουλών. Έχουμε ε, αυτούς τους τρεις άξονες που όμως πρέπει να σας πω να υπάρχει υποχρεωτική μείωση για τα κρατημέλη, να έχουμε κάποια μέτρα επί της τιμής και απαγόρευση εμπορίας. Οπότε για τα, το αποτέλεσμα ως ΓΚΟΕ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε Μάργκρετ Όκεν και η μείωση της ε, κατανάλωσης θα αλλάξει τον τρόπο ε, ε, που τα παίρνει ο κόσμος γιατί είδαμε ως ΓΚΟΕ ότι προωθήσαμε κάποια πιο αυστηρή νομοθεσία και μέσα σε τρία χρόνια είπαμε να μειωθεί κατά 50% η κατανάλωση και να φτάσει στο 100% σε τρία χρόνια. Και να έχουμε τέτοιες βιοαπικοδομήσιμες σακούλες για, για να μειωθεί η επικίνδυνοτητα τους. Οπότε έτσι βλέπουμε ότι προχωρούμε προς ε, πιο μακρές ε, προθεσμίες. είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να ε, υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν την εφαρμογή της νομοθεσίας με κοινή μέθοδο και υποέλεγχο της Κομισιόν. Και εν κατακλείδη θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν οι περιβαλλοντολόγοι και τα κινήματά τους σε αυτή την υπόθεση ούτως ώστε τελικά να έχουν μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Ριβασί για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τη συνάδελφό μου την οικολόγο, την Μάργαρετ Άουκεν που συνέγραψε αυτό το κείμενο για το Κοινοβούλιο και την ευχαριστώ και για την ποιότητα των διαπραγματεύσεων και για το επιτευχθέν αποτέλεσμα σήμερα θα ψηφίσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη μείωση των πλαστικών σακουλών εν ώψη τη υιοθέτηση του μέτρου από το Κοινοβούλιο. Πλαστικέ σακούλε πράγματι μέχρι τέσσερι αιώνε χρειάζονται για να διαλυθούν και ωκεανοί είναι γεμάτοι από τα μωριά του. Έχουν πολυθυλένη που παράγεται το πετρέλαιο και οι πλαστικέ σακούλε είναι πληγή για το περιβάλλον και όπω υπόθηκε πραγματικό δηλητήριο πρέπει να ληφθούν μέτρα ε, μεγάλη εμβελία για να μειωθεί αυτή η ρήπανση και αυτό είναι δεδομένο σήμερα, θα υπάρξει μία μείωση, καταναλώνουμε 200 σακούλες κατά κάτοικο, θα είναι 90 ε, μέχρι, σε, μέχρι 10 χρόνια. Και όταν... Λοιπόν, λοιπόν, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας και το οικοσύστημα και το νερό είναι στο επίκεντρο της προβληματικής που εξετάζουμε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο πέρα, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως λέμε στα γαλλικά. Ο, τις βιοδιασπόμενες, ε, οξυ, βιοδιασπόμενες σακούλες δεν είναι πραγματικά βιοδιασπόμενες, ε, διαλύονται σε μικρομόρια και αυξάνουν το κίνδυνο όσον αφορά το οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει, κύριε Πίτροπε, όταν θα, θα φάτε στρίδια αύριο μεθαύριο, σε αυτά τα στρίδια και στο νερό που περιέχουν θα βρείτε λοιπόν μικρομόρια. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προχωρήσει πιο πέρα απαγορεύοντας αυτό, ε, αυτές τις βιοδιασπόμενες ακούλες και δεν το έκανε Λοιπόν, προτιμήσατε να προστατεύσετε ιδιαίτερα συμφέροντα παρά να εμποδίσετε αυτή τη ρήπανση που θα επηρεάσει και θα πλήξει την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, για το EFTD, η κυρία Λανόρα Εύη για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φτάσαμε στην τελική φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ήταν πολύ δύσκολη από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εντυπωστήκαμε τα μάλα από, από τις ανησυχίες που δημιουργήθηκαν όταν διαβάζαμε τον αντίκτυπο των μέτρων. Κυρίως διαβάσαμε ότι ζημιά δημιούργησαν αυτές οι σακούλες στο περιβάλλον και κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όμως εξίσου εντυπωσιάστηκα βλέποντας τη σοβαρότητα και τον κατεπίγουσα ανάγκη αντιμετωπίσει του φαινομένου, το πώς ε, δεν είχε σαφείς στόχους η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι εύκολο αυτό που προσπαθούσε να πετύχει η κυρία Άουκεν. Ήθελε να έχει συγκεκριμένε προτάσει που θα κάνει και χάρη στη δουλειά τη έχουμε ένα κείμενο που είναι μεν ατελέ και βελτιώσιμο, όμω είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε, βλέποντα επίση και την, ε, πόσο αντιστάθηκε στη συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, η Ιταλική Αντιπροσωπεία τη ομάδα EFTD θα υποστηρίξει την πρόταση για, και την πρόταση αυτή και τη σύναψη συμφωνία με το Συμβούλιο. Τώρα από τους μη εγγυγραμμένους ο κύριος Τούκερ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σοφία της αποφάσισε να βάλει έναν επίτροπο για την καλύτερη νομοθεσία. Ο κύριος Τίμερμανς, ο αντιπρόεδρος. Η καλύτερη νομοθεσία λοιπόν είναι κάτι που χρειάζεται γιατί ο Ολλανδός ε, φορολογούμενος ε, έμεινε έκπληκτος ε, όταν άκουσε ότι ασχολείστε με το μήκος ε, της σκάλας, ε, τη, πόσο στραβές είναι οι μπανάνες και πόσο, πόσα ψωμάκια κανέλας πολλούνται. Με τον κύριο Τίμερ μας ήμασταν σύμφωνοι όταν ήθελε να καταργήσει την σακούλα αυτή και τις σχετικά, τις σχετικά μέτρα και σωστό αυτό, γιατί πρόκειται για ένα περτό μέτρο, αλλά τώρα τα πέταξε όλα αυτά στα σκουπίδια. Και ουσιαστικά είναι ο πιο καλός ε, και πιο καλοπληρωμένος μεταφραστής διερμηνέας του κυρίου Γιούγκερ, ο κύριος Τίμερμαντς. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή. Πολλές υποσχέσεις, αλλά ε, δεν ε, ανταποκρίνονται οι πράξεις. Ναι, λέει η Πρόεδρε, πολύ λυπάμαι, αλλά τελείωσε ο χρόνος ομιλίας σας. Διακόπτη Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πέτερ Λίζε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν για την εξέβρεση αυτή την ε, αυτό το συμβιβασμό για τις πλαστικές σακούλες γιατί να ευχαριστήσω και την Μαρία, κυρία Άουκον, την κυρία Όλβανη με πολύ μεγάλη εμπειρία από την εθνική πολιτική και από άλλους τομείς και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων από το ΕΛΚΑ. Έχουμε ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Στον ειρηνικό υπάρχει ένα πλαστικό χαλί με τρεις φορές το μέγεθος της Ευρικής Χερσονήσου. Το έχουμε συζητήσει αυτό σε διάφορες περιστάσεις. Ελπίζουμε η σημερινή νομοθεσία να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος και αυτό το ζω στις συζητήσεις με τους πολίτες. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και συμφωνεί με το γεγονός ότι ασχολούμαστε με αυτό. Έχουμε σαφείς διατάξεις για τη μείωση των πλαστικών σακούλων, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό επίσης να υπάρχουν, να επαφίεται στα κράτη-μέλη ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουν, να μην υπάρχει ευρωπαϊκή απαγόρευση. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα. Η Ιρλανδία και τα σκανδιναβικέ χώρε καταφέραν να το πετύχουν χωρί απαγορεύσει, αλλά με οικονομικά κίνητρα, με οικονομικά μέσα, τα οποία οδήγησαν σε δραματική μείωση των πλαστικών σακούλων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε, κατά πόσον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα της αγοράς και όχι απαγορεύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω βήματα και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επιτροπός Βέλα, αλλά και οι αντιπρόεδροι, οι αρμόδιοι θα έχουν υπόψη στο θέμα της πλαστικής σακούλας όταν θα μας υποβάλουν προτάσεις για την κυκλική οικονομία. Το φθινόπωρο. Γιατί και σε άλλα θέματα θα πρέπει να δούμε τι μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο στο θέμα της πλαστικής σακούλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λίζε, μία μπλε κάρτα από τον κύριο Τίμπο Σάνια. Έχετε... Την αποδέχεστε. Κύριε Σάνια, έχετε 30 δεύτερα στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Στην συζήτηση αυτή, διάφοροι συνάδελφοι όπως ο κύριος Ελίζα μας ε, ανέφεραν ε, ποιες είναι οι προσδοκίες στα κράτη-μέλη και τι ζητούν οι καταναλωτές. Εδώ όμω δεν μπορεί να μείνουμε σε επίπεδο γενικότητων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη μείωση τη κατανάλωση, Ποια μέτρα χρειάζεστε για να πετύχουμε τη μείωση αυτή. Ο κύριος Λίζε έχει 30 δεύτερα για την απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Συχνά μας ε, λένε ότι στα καταστήματα δεν θα πρέπει να ζητάμε πλαστικές σακούλες και πολλοί πολιτές απαντάνε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ναι, κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται. Νομίζω ότι μιλάνε εξ ονόματος του κόσμου. Στην Ιρλανδία, ωστόσο, έχει μπει ένα τέλος για τις ε, ελαφριές αυτές τις πλαστικές σακούλες άλλα συστήματα τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά από μια απαγόρευση. Εντυπωσιακά λοιπόν το αποτέλεσμα της Ιρλανδίας, χωρίς να υπάρχει απαγόρευση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτρο, ευχαριστώ. Αυτή η οδηγία που σήμερα θα εγκρίνουμε στο Κοινοβούλιο πάει πολύ παραπέρα από ένα απλό αποτελεσματικό εργαλείο. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν αρκεί για να σβήσει από τη μνήμη μα ε, τη φοβερή φωτογραφία ε, τη θάλασσα γεμάτη από σακούλε πλαστικέ. Κάθε σακούλα που πετάμε ε, κάνει 150 χρόνια να εξαφανιστεί. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Οπότε ε, ξεκίνησε εδώ και τόσα χρόνια αυτή η κατανάλωση και επομένως τώρα θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε την κυκλική οικονομία ως ε, οικονομικό μοντέλο. Πρόκειται για μια επανάσταση. Οπότε τώρα έχουμε αυτή την οδηγία. Είναι πάνω από ένα μέσον. Είναι ένα σύμβολο του πώς μπορεί κανείς να περάσει σε μια πιο βιώσιμη ε, κατανάλωση. Από την σχεδίαση μέχρι την κατανάλωση. Να έχουμε κάποια υλικά που σέβονται το περιβάλλον αναζήτηση κάποιων εναλλακτικών ίσως για ε, να ενθαρρυνθεί η, ε, η χρήση εκ νέου και η υπεύθυνη χρήση. Ε, αυτό αφορά στο πόσο χοντρές θα είναι, πόσο θα ζυγίζουν αυτές οι σακούλες και έτσι να κάνουμε αυτό το μετασχηματισμό, αυτή τη μετάβαση που θέλουμε και να δούμε τι γίνεται με τυχόν εναλλακτικά υλικά που να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα Έχουμε αυτό το στόχο λοιπόν του 2020 για 90 σακούλες ε, ανά άτομο κλπ. Και έτσι να έχουμε ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο να καταβάλουν προσπάθεια και οι άνθρωποι και οι χώρες. Και αξίζει για το βελτίο όλος ο πλανήτης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέτσελ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, τα αριθμητικά στοιχεία για τη μείωση τέτοια σακούλα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανησυχητικά και το γεγονό ε, που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο, για τον οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο μέλλον είναι σαφές. Έχουμε ε, άσκοπη σπατάλη της ενέργειας, ε, δεν έχουν καλό, καλή διαρκεία ζωής και μεγάλη βλάβη προξενού στο περιβάλλον. Και όλα αυτά μας οδηγούν για, σε μια σωστή ρύθμιση, σε σωστά μέτρα και όρια. Και γι' αυτό η προσέγγιση εδώ είναι απόλυτα σωστή. Για τη χρήση τέτοιων σακούλων με πάχος λιγότερο από 15 χιλιοστά. Αλλά το αποτέλεσμα ενδεχομένως να είναι αντιπαραγωγικό, γιατί ενδεχομένως να κάνουν πιο παχές τις σακούλες ε, η παραγωγή και έτσι θα, κατα... καταλάβουμε πιο πολύ ενέργεια και θα υπάρχει μεγαλύτερη ρήπανση στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπέρδρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο πάνω από 8 δισεκατομμύρια πλαστικέ σακούλες καταλήγουν στον απόβλητο στην Ευρώπη. Όχι μόνο αυτέ οι πλαστικέ σακούλες πλήττουν την ύπεθρο, αλλά και τα ποτάμια μα και οι θάλασσέ μα. Είναι θανατηφόρε για τα θαλασσοπούλια, τα ψάρια, τι φώκε, τα δελφίνια και άλλα, και στοιχεία τη έμβια ζωή. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω δράσεω ευρωπαϊκή. Μπορούμε δραματικά να περικόψουμε τη χρήση των σακουλών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση χρήση περίπου 200 ε, σακούλες κατά θα είναι και θα πάμε στις 40 μέχρι το 2025 κατά Τεράστιο βήμα προόδου, οπότε θα έχουμε καθαρότερους ωκεανούς και η πανίδα θα υποφέρει λιγότερο. Όμω επανειλημμένα οι συντηρητικοί ευρωβουλευτέ αρνήθηκαν να στηρίξουν αυτού του στόχου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι φιλελεύθεροι πολέμησαν στην κυβέρνηση κατά των συντηρητικών να εξασφαλίσουν ε, πέντε πένες ε, φόρος ε, κάθε πλαστική σακούλα που χρησιμοποιείται. Και εδώ οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές έδειξαν τα πραγματικά του χρώματα μην υποστηρίζοντας τα όρια που θέλει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που χρειάζονται. Αυτό δείχνουν ότι οι συντηρητικοί δεν θέλουν να προστατεύσουν πολύ το περιβάλλον. Η περικοπή της χρήσης των σακουλών θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πλε κάρτα έχετε. Δύο μπλε κάρτες. από την κυρία Γκέρλινγκ για 34. Με πρώτη εξ αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Μπέρντερ. Πιστεύετε ότι η πρόταση που έχουμε μπροστά μας είναι καλύτερη και θα είναι αποτελεσματικότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την πρόταση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου στηριζόμενη από τους φιλελευθέρους για την μείωση της χρήσης των πλαστικών σακουλών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Απάντηση. Ναι, η πρόταση αυτή είναι πανευρωπαϊκή πρόταση η οποία αφήνει στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ό,τι καλύτερο θεωρούν για την περιορισμό της Χρυσανακουλών στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους ε, φιλελευθέρους, το μανιφέστο τους. Ε, θέλαμε να επιβάλλουμε τις πέντε πένες σακούλα, σαν φόρο. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα αποτέλεσματα σε κάθε... Ε, έχετε και από την κυρία Ριβασί. Ε, από την κυρία Ριβασί, δεχόσαστε την άλλη ε, γαλάζια κάρτα, ναι. 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Μπέρντερ, είσαστε ευαίσθητοι για το περιβάλλον. Ποια είναι η θέση σας λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουμε απογορεύσει την χρήση των πλαστικών σακουλών των οξυγονοβιοδιασπομένων. Απαγορεύουμε αυτό που φαίνεται αλλά όχι αυτό που δεν φαίνεται διότι υπάρχουν διάφορα οικονομικά συμφέροντα. Απάντηση. Η χρήση των βιοδιασπομένων πλαστικών σακουλών είναι ένα πρόβλημα και δεν ε, λέω ότι το λύσαμε εδώ Α, τι συμβαίνει, αν οι βιδιασπόμενες όμως μπουν στον όλο κύκλο της βιοδιάσπασης ε, είναι επιβλαβής. Ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις βιοδιασπόμενες πλαστικές σακούλες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, για τα ψώνια, στις σακούλες που χρησιμοποιούν τα ψώνια. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Φλάνεγκαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο και συμφωνώ με την ιδέα του να υπάρξει κάποιο τέλος φόρος για να μειωθεί η χρήση των σακουλών. Αυτό έγινε στην Ιρλανδία και είχε αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και αντεπιχείρημα που να το λάβουμε υπόψη. Ποιο ήταν το, άλλο αποτέλεσμα. Έχουμε, αντί να έχουμε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, χρησιμοποιούμε ε, χάρτινες σακούλες έχουμε τώρα περισσότερη κατανάλωση, έχουμε περισσότερη κατανάλωση ύδατος ε, και δεν γίνεται ανακύκλωση. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπε κάποιο βουλευτή, ότι θα πρέπει να βρούμε ή να εφεύρουμε μια εναλλακτική. Ήδη ε, η εγγονή μου έχει την εναλλακτική λύση. Είναι μια σακούλα από λινάρι, από τέτοιο υλικό. Οπότε δεν χρειάζεται να εφευρουμε μια εναλλακτικη ηδη η εγγονη μου εχει την εναλλακτικη λυση ειναι μια σακουλα απο λιναρι απο τετοιο λιγο οποτε δεν χρειαζεται να επανεφευρουμε τον τροχό. Ούτε μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι που δεν το θέλουν. Με τον εξαναγκασμό θα οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα. Κάνει κάνει κάτι επειδή θέλει να το κάνει. Ας, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αφαιθούν τα κράτη-μέλη ελεύθερα να επιλέξουν. Βαλεντίνας Ματσουράνη, ένα λεπτό. Ποιτή συνάδελφοι, σε ένα λεπτό σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται ένα εκατομμύριο πλαστικές σακούλες και αυτό βλάπτει και την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν επιτάσσει γρήγορη αντίδραση. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, φιλόδοξοι και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να καταστεί οικονομικά ελκυστική. Κατά δεύτερον, πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μόνο αν οι στόχοι του κανονισμού έχουν τεκμηριωμένα αριθμητικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας τρόπος υπολογισμού και μόνο τότε να οριστούν δεσμευτικά μέτρα για την μείωση τρίτων ε, ένα διαφορετικό τέλος θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος αλλά να προσέξουμε προκειμένου να μην είναι ένα κρυφό τέλος αυτό το κόστος το οποίο θα ενταχθεί στην ε, τιμή παραγωγής. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθήσουμε αναλλακτικέ ε, μορφέ συσκευασία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Όμπερμαϊρ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα βλαβερέ ε, συνέπειες της πλαστικής σακούλας για το περιβάλλον. Καλωσορίζω λοιπόν τη σημερινή πρόταση. Ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν αποτελεί παρά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Φορολογία και η τιμολόγηση δεν μπορούν να αρκέσουν. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει θα πρέπει αυτό το πλαστικό να στο εγκαταλείψουμε εντελώς. Και στόχος μας θα πρέπει να είναι βιολογικά αποικοδομήσιμα υλικά. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτά τα υλικά συσκευασία ε, για φιάλες ε, και τα λοιπά μπορούν να μην χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ομάδες εργασίας και θα πρέπει όλα αυτά κυρίως να γίνονται σε πέτα κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιλάρα Γιούσο, για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτές οι σακούλες οι πλαστικές είναι πηγή πολλών προβλημάτων για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα κυρίως για τη θάλασσα. Και τα κράτη-μέλη κάναν μεγάλες προσπάθειες να μειώσουν την χρήση αυτών. Πολλά κράτη-μέλη πήραν κάποια μέτρα. Και με αυτή την οδηγία τώρα τα κράτη-μέλη θα έχουν διάφορα μέσα ούτως ώστε να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους σκουπίδια, να μην χρησιμοποιούνται αυτές οι σακούλες χωρίς να χρειάζεται. Γι' αυτό γίνεται στη χώρα μου ε, σε σούπερ μάρκετ και φαίνεται κάποια αποτελέσματα και να έχουμε και εξαιρέσεις για κάποιες λεπτές σακούλες που χρειάζονται ε, πολλές φορές για την αγορά ε, σε επίπεδο χονδρικής κάποιων ε, τροφίμων ε, και κάποιων ζωοτροφών οπότε θα πρέπει επομένως να κάτσουμε και να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά της κάθε εναλλακτικής λύσης θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια αλλά και στους σκιώδεις εισηγητές οι επίσης απέσπασαν κάποια αξιόλογα αποτελέσματα μετά από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Νομίζω ότι το κείμενο θα υιοθετηθεί, θα, θα εγκριθεί με ευρεία συνένεση. Η κυρία Κάντενμαχα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συχνά ως βουλευτές αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα να ε, εξηγήσουμε τις αποφάσεις μας στο ευρύ κοινό. Και αυτό πολύ απλά επειδή έχουμε μια μεγάλη επιθυμία στην οποία αντιποκρινόμαστε των Ευρωπαίων. Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων είναι υπέρ της μείωσης της πλημμυρίδας αυτής πλαστικού. Και στην Αυστρία, 73% του κόσμου τάχθηκε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης. Κάνουμε λοιπόν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή για τη μείωση σε πρώτη φάση και για την ευαισθητοποίηση γιατί σήμερα απαρίσκεπτε παίρνουμε τις σακούλες αυτές. Και σας καλώ όλους να μην πετάτε για κάποιο διάστημα αυτές τις σακούλες, αλλά να τις μαζεύετε, να δείτε τι βουνό θα φτιάξετε σε σύντομο χρονικό διάστημα. 400 χρόνια λοιπόν χρειάζεται αυτό το βουνό σακούλων για να διασπαστεί. Αυτό γιατί για 20-30 λεπτά άνεσης μέχρι να πάμε στο σπίτι μας. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξουν ευέλικτες ρυθμίσεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ διαφορετικό το τοπίο 200-400 σακούλες ανά Ευρωπαίο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Εγώ έχω να πω ότι θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις από πλευράς των πολιτών για τη μείωση αυτών των σακουλών. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Τζέιμ Νίκολσον τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα εργασιών το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε πει ο κύριος Ζαν Κλοντ Γιούγκερ ότι ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη για μεγάλα θέματα και μικρότερη για πιο μέτρια πράγματα και μικρά πράγματα. Η οδηγία φοβάμαι, αυτή που συζητούμε είναι ένα παράδειγμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερβολικά μεγάλη και υπερβολικά φιλόδοξη όσον αφορά μικρά θέματα. Σαν ένα θέμα που χρησιμοποιείται καθημερινά στα νοικοκυριά στην Ευρώπη, η πλαστική σακούλα δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερη, Ποια είναι η βασική αρχή για τη μείωση της βλάβης των περιβάλλων από τις πλαστικές σακούλες. Ε, είναι ένας στόχος που μπορούμε όλοι να στηρίξουμε, να μειωθεί η χρήση. Αλλά τα μέτρα της συμφωνίας της δεύτερης ανάγνωσης ίσως να είναι πολύ περιοριστικά και ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστούν. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ όσον αφορά την κατανάλωση μεταξύ των κρατών μελών σε αυτά σακούλε. Στην εκλογική μου περιφέρεια μειώσαμε τι πλαστικέ σακούλε κατά 72%. Διότι επιβάλαμε ένα τέλος πέντε πενών. Ε, αφήστε το θέμα να το ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη, είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίση, η οποία επίση έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε. Κάποια στοιχεία αρκούν παρά. Λοιπόν, πέντε δευτερόλεπτα χρειάζεται για να χρησιμοποιηθούν, πέντε λεπτά για να χρησιμοποιηθούν σακούλες και 500 χρόνια για να αποσυντεθούν. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντικό συμβιβασμό που έχει πετύχει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να αποθαρρυνθεί η χρήση του. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη θα έχουν την επιλογή να μειώσουν τον αριθμό των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται κατά άτομο κάθε χρόνο, όχι πάντα από 45 μέχρι το 2025 και να μειωθεί η χορήγηση μέσω των καταστημάτων μέχρι το 2018 είναι λογικό. Δυστυχώ, βλέποντα τι διαφορέ που υπάρχουν στην Ευρώπη, τέσσερι πλαστικέ σακούλε καταναλωτή κατά το χρόνο στη Φιλανδία, 400 στην Πολωνία, στην Πορτογαλία. Ε, ε, λοιπόν, δεν είναι βιώσιμη όλη η προσέγγιση. Λοιπόν, δέκα χρόνια έχουμε στη διάθεσή μα για να ε, ακολουθήσουμε του καλύτερου μαθητέ στην τάξη. Μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα η Ευρώπη, πρέπει να το κάνει αυτό. Μιλάμε για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να εμπνευστούν από τι βέτε πρακτικέ του Βορρά, όχι μόνο από τον Βορρά και από αλλού. Ε, στην Ιρλανδία είναι το κάτω του Λουξεμβούργου. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Επίση ε, για ένα λεπτό, κύριο Πέταμαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταθέσω μία τροπολογία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναπαιμφθεί αυτή η τροπολογία σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης πλαστικής σακούλας στα καταστήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει οι ίδιοι άνθρωποι μόνοι τους να αποφασίζουν τι ακριβώς επιτιμούν να χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν τα ψώνια τους. Και μην υποτιμάτε τους ανθρώπους. Όταν κάτι είναι λογικό, το αποφασίζουν μόνοι τους. Και όταν ε, χρειάζονται ε, κάτι για να τυλίξουν ε, τα ψώνια τους, ε, κρίνουν μόνοι τους αν θέλουν να είναι χαρτί ή πλαστικό. Εάν επιβάλλουμε αυτή την απαγόρευση, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν περισσότερες μικρές πλαστικές σακούλες. Θα τους ε, οδηγήσουμε στο να χρησιμοποιούν πλαστικά φύλλα ε, για να τυλίξουν τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι όσοι επιθυμούν να απαγορεύσουν την πλαστική σακούλα ε, ποτέ δεν την έχουν χρησιμοποιήσει γιατί νομίζω ότι εκείνοι που λένε ότι θέλουν να τα απαγορεύσουν είναι απλά υποκριτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Jean-François Σάικ επίσης για ένα λεπτό. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν κοιτάξουμε επιφανειακά το κείμενο αυτό, που λέει να μειώσουμε την κατανάλωση λεπτών πλαστικών σακουλών θα έπρεπε να μας βρίσκει σύμφωνος, ομόφωνα. Όμως, αν το κοιτάξουμε πιο κοντά, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό, ένα φάτα μοργάνα στο οποίο μας έχει συνηθίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε μια λεπτομέρεια για να μην αμφισβητήσουμε το ίδιο το σύστημα. Προωθούμε μια διακοσμητική οδηγία για τις σακούλες αυτές, ενώ από την άλλη μεριά ενθαρρύνουμε περισσότερες μεταφορές και περισσότερη αλληλεξάρτηση διεθνώς. Η πολιτική αποτελεσματικότητα και η οικολογική στάση αυτού του κειμένου είναι κάτι πολύ αμφισβητήσιμο. Διότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε ένα μικρό δείγμα μόνο συσκευασία. Έτσι λοιπόν απαγορεύουμε αυτές τις σακούλες, ενώ από την άλλη μεριά ενθαρρύνουμε τον πολλαπλασιασμό άλλων συσκευασιών. Από την άλλη μεριά οι λαοί αναγκάζονται να δεχτούν ένα νέο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα εμβληματικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομοθετικό κείμενο που δεν είναι σωστό. Κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο πια, οι πλαστικές σακούλες που συμβολίζουν την κοινωνία της κατανάλωσης. Είναι πολύ καλό που έχουμε επιτέλους συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δείχνει περισσότερη ευαισθησία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα ρητό των Ινδιάνων που λένε ότι τη γη αυτή την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή τη γη. Οι πλαστικές σακούλες αναμφίβολα αποτελούν τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια θετική οδηγία και τα κράτη-μέλη πρέπει να την ε, εφαρμόσουν. Εξάλλου, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν το στόχο. Προτιμάω κίνητρα για την απαγόρευση. Σε σκανδιναβικές χώρες, στην Ελλαδία και αλλού έχουμε τέτοια παραδείγματα όπου τα κίνητρα φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την Κροατία, ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ποτάμια μας και η αδριατική μας θάλασσα. Πολλές φορές το έχω πει ότι έχουμε πρόβλημα με τις πλαστικές σακούλες οι οποίες φτάνουν σε μας από την Αλβανία στα κρατικά ύδατα και τις ακτές μας με φορτηγά πλοία είναι κάτι το οποίο καταστρέφει την οικονομία μας, τον τουρισμό μας και φυσικά το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συζητήσουμε αυτό το θέμα και με τις χώρες που δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπλε κάρτα έχετε από τον κύριο Γιάνκοτσης. Δέχεστε. Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα κύριε Γιάνκοτσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Σούσα που δεχτήκατε την μπλε μου κάρτα. Θέλω να να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα της διασυνοριακής ρήπανσης. Από την Αλβανία ε, λέτε και από τον Έρετβα το ποτάμι, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για την προσχώρησή τους θα έπρεπε να θέσει αυτή την προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν περισσότερο οι διαπραγματεύσεις. Προσχώρηση των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάκοβιτς που θέτετε αυτό το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι η Αδριατική θάλασσα είναι κλειστή θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλες οι χώρες οι οποίες βρίσκονται γύρω από την θάλασσα αυτή να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Όμως οι χώρες αυτές δεν είναι όλες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία, η Βοσνία Ζεγοβίνη για παράδειγμα ή το Μαυροβούνιο. Οπότε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εγώ έθεσα επανειλημμένο στο ζήτημα αυτό. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα κεφάλαια τα οποία ε, διαπραγματευόμαστε με νέες χώρες προς προσχώρηση. αλλιώ. δεν θα μπορούμε να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ένα, 1,5 λεπτό η κυρία Πόλτου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, όσον αφορά τις ε, πλαστικές σακούλες ε, πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το σκέφτονται, απλά χρησιμοποιούν αυτές τις σακούλες και νομίζω ότι υπάρχει στο σπίτι καθενός από εμάς ένα συρτάριο που έχουμε αυτές τις σακούλες και τις χρησιμοποιούμε κατά καιρού. Την επόμενη φορά όμως που θα δείτε κάποιον να πετάει μια πλαστική σακούλα στη θάλασσα ενώ εσείς ε, κάνετε ηλιοθεραπεία, μην ξεχνάτε ότι θα μπορούσατε κάτι να έχετε κάνει γι' αυτό. Ο αριθμός της ε, πλαστικής σακούλας ε, που τελικά καταλήγει στις θάλασσες είναι τραγικός. Και αυτό το γεγονός νομίζω ότι και μόνο το αρκεί για να περιορίσουμε τις πλαστικές σακούλες στο έγγραφο αυτό ε, περιγράφονται πιθανές λύσεις ε, στο πρόβλημα. Η χώρα από την οποία προέρχομαι εγώ δεν ε, παρουσιάζει υψηλή κατανάλωση πλαστικής σακούλας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χαιρόμαστε το να υπάρχει η δυνατότητα στις χώρες να αποφασίζουν μόνες τους. Τα κράτη-μέλη βεβαίως μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους πώς μπορούν να επιτύχουν το στόχο τους και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να προσαρμόσουν τις ε, λύσεις στις ε, ιδιαιτερότητες τους. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε την πλαστική σακούλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκέρεκε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί ερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδα τρεις ε, πλαστικές σακούλες ε, που ήταν στο ποτάμι. Ε, μηδέν λοιπόν ανακύκλωση και μηδέν φροντίδα για το περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι πλέον παγκόσμιο εδώ και αρκετό καιρό και δεν μπορούμε να το συγκαλύπτουμε. Θέλω λοιπόν το διευκνήσω. Μιλάμε για κάτω εκατοντάδες χιλιάδες τόνους πλαστικού που ε, ρηπαίνουν τις ε, θάλασσες πολλά απόβλητα κάθε χρόνο έχουμε και προστίθενται άλλα 13 εκατομμύρια τόνους. Ε, πολλοί μιλάνε για την 7η Ήπειρο, 3,4 ε, χιλιάδες χιλιόμετρα στην, ανάμεσα στην, στην, Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια και την ε, Χαβάη. Και όλα αυτά είναι το σύνολο της πλαστικής σακούλας. Στα παιδιά μου τους λέω ότι αυτές τις πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούν. Το ίδιο όμως ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Ευτυχώς λοιπόν που αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα στην Ευρώπη. Το καθήκον μας πρέπει να είναι να ανακυκλώνουμε τις σακούλες και αν το καταφέρουμε αυτό θα κατακτήσουμε την 7η Ήπειρο και θα ελαφρύνουμε, ε, θα απαλύνουμε ε, τον κόσμο από αυτό το δεινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπάλτσοφ, επόμενος ομιλητής, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η πρακτική χρήση αυτών των σακουλών έχει αποδειχθεί καταστροφική. No... Σα διακόπτω διότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Παρακαλώ, ξανά ξεκινώ. υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Μήπως μπορεί η γερμανική καμπίνα να ξαναμιλήσει. Η χρήση των πλαστικών σακουλών είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλα τα κράτη-μέλη με τεράστιο αντίκτυπο. 8 δισεκατομμύρια σακούλες πηγαίνουν στις χωματερές κάθε χρόνο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Είμαι υπέρ του κανονισμού, αν και, και μέσω μιας οδηγίας θα μπορούσαν τα κρατημέλη να μεταφέρουν τις διατάξεις αυτές στις εσωτερικές ένομες τάξεις. Έτσι θα υπήρχε περισσότερη ευελιξία προς την εφαρμογή. Πρέπει επίσης να ρυθμίσουμε την ψευδή σήμανση. Δεν είναι όλες οι σακούλες ε, βιοδιασπόμενες. Πολλές φορές η σημαντική αυτή είναι παραπλανητική διότι αφορά μόνο την διάσπαση σε πολύ μικρότερα τεμάχια. Θέλουμε πραγματικά λιπασματοποιήσιμες σακούλες και όχι απλώς διασπόμενες σε μικρότερα κομμάτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Φαντσέσκο Κάμπους για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μιλάμε για την κατανάλωση πλαστικών σακουλών, μιλάμε για το περιβάλλον μας. Θέλουμε να νομοθετήσουμε για να έχουν καλύτερη ζωή τα παιδιά μας. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και όμως πρόκειται για εκατομμύρια Ευρωπαίους που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Μετά από τρία χρόνια μάχης καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για να μειωθούν οι σακούλες αυτές. Σημαντική συμφωνία και σημαντική για να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας. Όπως λέει η εκστρατεία ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το είπαμε εδώ και σήμερα, πέντε λεφτά χρειάζονται για να κατασκευαστεί μια τέτοια σακούλα. Πέντε λεπτά θα τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα εξαφανιστεί μετά από 50 χρόνια. Επειδή διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα, νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, η απόφαση που πήραμε, δηλαδή σε 40 σακούλες ανάτομο το 2025 να μειωθούν οι σακούλες αυτές και να αποφασίσει το κάθε κράτος πώς. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί για να γίνει αλλαγή στην οτροπία. Αυτό είναι που χρειάζεται. Και συμφωνώ με τον κύριο Φλάνακαν. Οι, οι γιαγιάδες μας θα μπορούσαν να μας δώσουν μεγάλα μαθήματα. Στην Καταλωνία προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο από το 2007. Και έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι όντως 54% θα έχουμε μειώσει μέχρι το 2020 την κατανάλωση σακουλών ανά άτομο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια την κυρία Όκεν για το έργο της. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάμπους. Ε, κύριε Γκάμπους υπάρχει μια μπλε κάρτα ε, για σας από τον κύριο Γκόνης Γρούπε. Τι δέχεστε αυτή την μπλε κάρτα. Παρακαλώ έχετε 30 ε, δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Πρέπει να βρούμε τρόπο για να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών σακουλών. Για μένα ο μόνος τρόπος είναι να σταματήσουμε την δωρεάν διάθεσή τους. Δεν πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν και η πιο αποτελεσματική λύση. Και πότε θα αρχίσουμε να χρεώνουμε αυτές τις σακούλες το 16-18, τι πιστεύετε. κύριος Το να τις χρόνουμε είναι μια εναλλακτική λύση, αλλά καλύτερη εναλλακτική είναι αυτή που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να αλλάξουν νοοτροπία κάθε φορά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια πλαστική σακούλα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γιόρλα, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Βέλα. Ε, είσαστε αρμόδιους ε, και για τη θαλάσσια πολιτική και το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι πολλές από τις ε, πλαστικές σακούλες καταλήγουν τελικά στις θάλασσες, στους ποταμούς και έχουμε λοιπόν αυτά τα τεράστια ε, χαλιά αποβλήτων στους ωκεανούς. Ε, ένας συνάδελφος μίλησε μάλιστα για την 7η Ήπειρο. Γνωρίζουμε ότι αυτό το πλαστικό υλικό έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Ε, είναι και διαβολικό γιατί τα ψάρια πιστεύουν ότι είναι τροφή, τα καταπίνουν και μετά είτε αρρωσταίνουν είτε πεθαίνουν. Άρα δηλαδή επιγόντως κάτι πρέπει να γίνει για να περιοριστεί αυτή η πλημμυρίδα της πλαστικής σακούλας. Και επιπλέον και εγώ πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να μοιράζονται δωρεάν οι πλαστικές σακούλες. Θα πρέπει κανείς να πληρώσει αν θέλει να έχει πλαστική σακούλα εφόσον ε, τη χρειάζεται. Και υπάρχουν και δυνατότητες ε, να παγορεύσουμε ε, τις ε, πλαστικές σακούλες γιατί υπάρχουν αλλακτικέ λύσεις ε, και σε άλλα θέματα απαγορεύουμε τις χειρότερες μεθόδους και με τον τρόπο αυτό προάγουμε τις καλύτερες. Ευχαριστώ την κυρία Άουκεν η οποία παρέμεινε πιστή στους στόχους του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν ήταν εύκολο στο πλαίσιο της τριμερούς συζήτησης. Η Κομισιόν μάλιστα ήθελε να αποσύρει την πρότασή της. Είναι λοιπόν πολύ καλό που έχουμε ένα καλό νόμο και κύριε Μπέλα, κύριε Επίτροπε, η δική σα δουλειά είναι να εφαρμόσετε το νόμο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ ο ε, κύριος Κάμπλ Μπάνεμαν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, πολλές ε, συζητήσεις ε, έγιναν ε, σχετικά με τις σακούλες αυτές και με την καινούργια τεχνολογία η οποία όπως σας είπα έχει συμβάλει πάρα πολύ ε, στη μάχη κατά της σακούλας. Ε, αυτή λοιπόν η καινοτόμος ε, τεχνολογία έχει προχθεί από μια εταιρεία στην Ανατολική Εγκλαία με πάρα πολλούς, 30 περίπου υπαλλήλους που είναι πολύ αφοσιωμένοι. Εγώ τους αποτείω φόρο τιμής και νομίζω πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός στο μέλλον. Αυτή η τεχνολογία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ο εισηγητής έχει βέβαια ε, και κάποια συμφέροντα τα οποία επισημαίνει. Ο στόχος είναι βέβαια στην περίπτωση αυτή να εξαλειφθεί ένας ανταγωνιστής από την αγορά. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και χάρη τη δουλειά που έγινε από του συναντέλφου, του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ, οι Κομισιόν και τα Συμβούλια έδειξαν λογική και τέλο ε, απαγορεύεται αυτή η όξο βιοαπικοδομήσιμη τεχνολογία για τι πλαστικέ σακούλε. Κατόπιν τούτου θεωρώ θα πρέπει λιγάκι να περιμένουμε και να μην σπέβδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κάμπλ Μπένεμεν. Ε, δύο μάλιστα μπλε κάρτε ε, για εσά. Ε, από τον Αγγενιού, κύριο Αγγενιού και από την κυρία Άουκεν. Δέχεστε και τις δύο μπλε κάρτες, παρακαλώ. Ο κύριος Αγγενιού είναι ο πρώτος. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε, αυτό είναι ασυνήθιστο. Είναι μια φιλική ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί και εγώ εκπροσωπώ την ίδια εκλογική περιφέρεια όπως ο προλαλή σα και ε, δεν νομίζω θα μπορούσα να μιλήσω στη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ Γι' αυτό λοιπόν ε, να πω λίγα πράγματα ε, περισσότερα για το ότι συμφωνούμε απόλυτα και οι δυο μας. Δεν είναι λοιπόν μάλλον σπάνιο να στηρίζει κάποιος ε, τον συνάδελφό του. Ναι λέει η πρώτη. Εντάξει ασυνήθιστο είναι αλλά οι μπλε κάρτες είναι για να γίνονται ερωτήσεις. Εσείς δεν κάνατε ερώτηση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κυρία, στην κυρία Άουκεν και μετά έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Ε, Πρόεδρε, εδώ βλέπουμε ε, ποιο είναι το πρόβλημα με τις όξο βιοαπικοδομήσιμες σακούλες. Είναι το πρόβλημα μιας βρετανικής εταιρείας. Εμείς δεν θέλαμε τη διάσπαση. Εμείς έχουμε αποδείξεις ότι οι όξο βιοαπικοδομήσιμες είναι χειρότερες από το τίποτα μάλιστα. Ε, θέλουμε τώρα η Επιτροπή να κάνει κάποια έρευνα και θέλω να ρωτήσω το συνάδελφό μου, εσείς τελικά είσαστε υπέρ του να γίνει μια έρευνα και αν αποδειχθεί ότι αυτές οι σακούλες είναι χειρότερες από τις κανονικές, τότε ελπίζω να μας βοηθήσετε να τις ξεφορταθούμε. Ο κύριος Κάμπλι Μπάνεμαν, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εγώ εκείνο που ζητάω είναι να υπάρχει μία τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη και να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Γιατί είμαι πεπισμένο και το ξέρω και από την εκλογική μου περιφέρεια ότι αυτή είναι μια πολύ καλή τεχνολογία η οποία θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ρήπανση. Λυπάμαι, αλλά υπάρχει κατάχρηση σε επιστημονικό πεδίο, ε, εκτοξεύονται επιθέσει εναντί σε αυτήν την εταιρεία. Α δούμε λοιπόν τα γεγονότα και α μην παραμένουμε πιστοί σε προκαταλήψει. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα παρακαλώ ο Φουντούλη για ένα λεπτό. Και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα για τι πλαστικέ σακούλες μεταφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα περιοριστεί η χρήση του, η οποία έχει επιφέρει μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. αρχικά θεωρούμε βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση την παρούσα έκθεση το οποίο όμω δυστυχώ δεν αρκεί. ειδικά στο θέμα των αποκαλούμενων ω αυτοδιασπόμενων πλαστικών σακουλών θεωρώ πω τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε είναι ανεπαρκή. ορισμένοι θησάβρισαν επειδή προωθούσαν το υλικό ω δίθεν φιλικό προ το περιβάλλον την ίδια ώρα που προκαλούσαν τρομερή οικολογική ζημιά. πιστεύω λοιπόν πως πρέπει να προτείνουμε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους. άποψή μου είναι πως πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης λεπτών και πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών κρατώντας μόνο εκείνες που έχουν αρκετό πάχος ώστε να είναι επαναχρησιμοποιούμενες και μάλιστα ο καταναλωτής να καταβάλει αντίτιμο για την απόκτησή τους πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες χώρες της ένωσης. όσον αφορά την αντικατάστασή τους πρέπει να επιστρέψουμε στη χρήση χάρτινων αποκλειστικά δε ανακυκλώσιμων. πιθανότατα αυτό να μην είναι ούτε τόσο βολικό ούτε συμφέρον οικονομικά όμως πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και θυσίες για την προστασία του περιβάλλοντος διότι οι μελλοντικές συνέπειες θα είναι καταστροφικές για ολόκληρο τον πλανήτη αν εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τη σημερινή πρακτική. ευχαριστώ. Επόμενη, κυρία Λουκατσέψκα, έχει το λεπτό για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία αυτή είναι μια θεραπεία. Παρά κάποιες διαφορές που υπάρχουν εδώ στο σώμα, οι πολιτικές ομάδες τη στηρίζουν. Όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους περισσότερους από τους προλαλήσαντες που είπαν πόσες πολλές σακούλες, εκατομμύρια σακούλες ρηπαίνουν το περιβάλλον και πόσο πολλά χρόνια χρειάζονται για να εξαφανιστούν. Να απορροφηθούν από το περιβάλλον. Το θέμα της ρήπανση λοιπόν και καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα και την πανίδα είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι κάποιες χώρες μέλη ήδη έχουν εισαγάγει μέτρα και έχουν την υποχρέωση να χρεώνουν τις πλαστικές αυτές σακούλες αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Χαίρομαι επίσης που βλέπω ότι η οδηγία αυτή δίνει τα μέσα που χρειάζονται οι χώρες μέλη προκειμένου να πετύχουν τους στόχους αυτούς και ελπίζω να φανούν φιλόδοξα στην επιτευξή του. Η τιμή τώρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις κοινωνίες. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, στις οικογένειες, ε, στα σχολεία να μαθαίνουν τα παιδιά τις επιπτώσεις που έχουν οι σακούλες αυτές στο περιβάλλον. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό των παιδιών, να το καταλαβαίνουν τι σημαίνει η βιοαποδομήσιμη συσκευασία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Ανδρουλάκης, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Υπολογίζεται ότι το 2010 99 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες χρησιμοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το νούμερο μεταφράζεται σε 200 σακούλες ανά άτομο. Η πλειοψηφία αυτών είναι οι λεγόμενες λεπτές πλαστικές σακούλες, τις οποίες τις βλέπουμε κυρίως στα σούπερ μάρκετ και στα εμπορικά καταστήματα. Έχοντας υπόψη ότι τις περισσότερες φορές οι σακούλες αυτές δεν ξαναχρησιμοποιούνται. Η επιβάρηση του περιβάλλοντος είναι σημαντική ιδιαίτερα στα υδάτινα οικοσυστήματα. με την παρούσα οδηγία γίνονται οι απαραίτητε τροποποιήσει στην νομοθεσία για τα απόβλητα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειε προ το περιβάλλον. το κοινοβούλιο ζητούσε από την αρχή να μπουν συγκεκριμένοι στόχοι μείωση και τη χρήση τη λεπτή πλαστική σακούλα. με τη συμφωνία που επετέφθη, τα κράτη μέλη έχουν δύο επιλογέ μπορούν είτε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση στου 90 ανά άτομο μέχρι τέλος του και στις 40 μέχρι το τέλος του 2025. Είτε να απαγορεύσουν ως δεύτερη επιλογή την παροχή τους στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων και προϊόντων το αργότερο ως το τέλος του 2018. Καλωσορίζω και στηρίζω τη συμφωνία αυτή και πιστεύω πως βάζουμε σήμερα τις βάσεις για την αντιμετώπιση μιας πολύ σημαντικής πηγής μόλυνσης. Ρενάτε Μπριάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την κυκλική οικονομία και ε, κάνουμε ένα σημαντικό πήμα προς ε, για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας. Τα κράτη-μέλη έχουν ακριβείς ε, κανόνες. Πέρυσι η Ιταλία εισήγαγε την απαγόρευση της δωρεάν πλαστικής σακούλα αλλά αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους στο πλαίσιο των πολιτικών της πρόληψης διαχείρισης ε, των αποβλήτων, υπάρχουν τα σωστά εργαλεία της ε, διαχείρισης ε, και της βιομηχανικής έρευνας. Η διανομή της πλαστικής σακούλας είναι καταστροφική, κυρίως σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Μαζεύονται πάρα πολλά σκουπίδια και έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί στον Ειρηνικό κιανό ένα τεράστιο χαλί από πλαστικές σακούλες. Μιλάμε για δύο ή τρεις φορές το μέγεθος της Ιταλίας. Είναι απαραίτητο να δράσουμε ταχύτερα. Αυτό είναι δέσμευση γιατί μην ξεχνάμε τα παιδιά έχουν στραμμένα τα μάτια τους προς εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν θα δεχτώ πλέον ε, άλλη μπλε κάρτα από ανθρώπους ε, που έχουν ε, ήδη χρησιμοποιήσει το δικαίωμα. Πρέπει πια να προχωρήσουμε να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Δέκα έχουν ζητήσει το λόγο. Θα πάρω όμως έναν από κάθε πολιτική ομάδα. Ο πρώτος είναι ο κύριος Τζοβάνι Λαβία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της ε, τριμερού συνάντησης που είχα την ευκαιρία να προεδρεύω μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κατορθώσαμε με την εισηγήτρια και με το Συμβουλίο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Διακόπτη η πρόεδρος, πάλι δεν υπάρχει μετάφραση στα γερμανικά. Λυπάμαι, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Κύριε Επίτροπε, αυτή ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Κοινοβουλίου. Γιατί στο τριμερείς συζητήσεις με την εισηγήτρια και με το Συμβούλιο καταλήξαμε σε συμφωνία και όχι μόνο λειτουργήσε και διευκόλυνε η Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή τελικά που απέσυρε τη δική της πρόταση και απέμεινε η δικιά μας και με τον τρόπο αυτό στο τέλος του κειμένου έγιναν κάποιες παρατηρήσεις από την Επιτροπή σχετικά με την ατότητα εφαρμογή του κανονισμού. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία που την πέτυχαν οι συνομοθέτες ακριβώς όπως προβλέπετε από την κείμενη συμφωνία της ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνες. Θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Υπάρχουν λύσεις, έχουν υιοθετηθεί από κάποια κράτη-μέλη. Σήμερα λοιπόν έχουμε στόχο ε, σχετικά με την πλαστική σακούλα, έχουμε νέες ε, τεχνολογίες, γι' αυτό λοιπόν ας απαγορεύσουμε και ας απομακρύνουμε εκείνο που μοιάζει ότι δεν είναι το καλύτερο για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Νίκολα Καπούτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Η μείωση κατανάλωσης πλαστικής σακούλας ε, και λεπτής πλαστικής σακούλας ε, είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι πρωταρχικός. Ε, κυρίως μην ξεχνάμε ότι το 2010 πιστεύαμε ότι κάθε πολίτης χρησιμοποιούσε πολλές σακούλες, κυρίως ελευρές σακούλες. Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Κοινοβουλίο και συγχαίρω την κυρία Άουκεν για την πολύ καλή δουλειά δουλειά είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αρχική πρόταση Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστεί, να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η πλαστική σακούλα. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την κοινοτική νομοθεσία. Το κείμενο ε, προβλέπει και τη δέσμευση των κρατών μελών να παρουσιάζουν κάθε χρόνο μία αναφορά σχετικά με τη χρήση ελαφριάς ε, πραστικής ε, σακούλας. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν πιο αυστηρές δεσμεύσεις και κατόπιν τούτου θα υπάρχουν και συγκεκριμένα εργαλεία στα χέρια των κρατών μελών για να ελέγχουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ντεμεσμάκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε τι καταστροφή έχουμε στις θάλασσές μας. Αρκεί αυτό για να καταλάβουμε τη ζημιά που κάνουν αυτές οι πλαστικές σακούλες. Γι' αυτό και πρέπει να τις περιορίσουμε. Βέβαια, οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη είναι τεράστιες. Στη Φλάνδρα έχουμε καλά αποτελέσματα. Από το 2003 η χρήση των πλαστικών σακουλών έχουν μειωθεί κατά 80% και πάντα υπάρχει βέβαια περιθώριο ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται να υπάρξει μείωση εφόσον υπάρξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και εφόσον υπάρξει προστασία του περιβάλλον όλους τους πολίτες. Χρειάζεται βέβαια και ευελιξία να προσφέρουμε στις χώρες μέλη. Αυτή η οδηγία πιστεύω όμως ότι οδηγεί σε κάποιο λογισμό. Γιατί χρειάζεται κάτι πιο γενικό. Το πακέτο αυτό πρέπει να συνοδευτεί με διαρθρωτικά μέτρα πιο συγκεκριμένα, ώστε η οικονομία μας να μην πληγεί από τέτοιου τους μέτρα. Και εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριος Ιβαν Γιακοπτσίτς για ένα λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Εμείς Είμαστε μικροί καταναλωτέ τέτοιων ε, σεκουλών, κατά κεφαλήν. Ιδιαίτερα σε σύγκριση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Παρ' όλα αυτά, η Κροατία είναι σημαντικός παραγωγός τέτοιων σεκουλών και αυτό είναι πρόβλημα για μας, διότι κινδυνεύουμε να χάσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό προκαλεί με τη σειρά του άλλα προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι έχω εργαστεί σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο αλλά δεν είμαι εδώ για να υπερμηνθώ των συμφερόντων αυτού του κλάδου ίσα ίσα. Θεωρώ ότι οι σακούλες αυτές αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και τονίζω ότι αντιμετωπίζουμε στην Αδριατική ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσμα ακριβώς της διασυνοριακής ρήπανσης, πλαστικέ σακούλε που προέρχονται από την Αλβανία και ούτω καθεξής. Πρέπει και αυτό να μπει στη διαπραγματεύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ομιλητής ο κύριο Ιγκό Σούλτε ε, για ένα λεπτό. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Άουκεν, ε, για την έκθεσή της. Η έκθεσή της είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οι πλαστικές σακούλες Ε, χρησιμοποιούνται ευρέως και τα μέτρα τα οποία προβλέπει η οδηγία, τα μέτρα αυτά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Όμως ε, πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι αν οι καταναλωτές γνώριζαν ε, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ε, πλαστικής σακούλας, θα σκεπτόντουσαν διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να τους πούμε την αλήθεια για αυτές τις πλαστικές σακούλες. Βεβαίως οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Το 90% της πλαστικής σακούλας χρησιμοποιείται μία μόνο φορά και αυτό έχει ως συνέπεια το ότι αυξάνονται συνεχώς τα σκουπίδια. Κάθε χώρα λοιπόν οφείλει να κάνει προεκλογική εκστρατεία, ε, το πλαστικό ε, είναι ε, αρνητικό, δεν είναι καλό για την οικονομία και γι' αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Πολύ ωραία, λέει η πρόεδρος. Φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου Catch the Eye και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μπέλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και τα επικοδομητικά σχόλια. Αναφέρθηκαν παραδείγματα από κρατημέλη τα οποία έλαβαν μέτρα για να μειώσουν την χρήση τέτοιων σακουλών. Αυτά αποδεικνύουν ακριβώς ότι η δράση είναι αποτελεσματική. Κυρία Οκέν, Ανέφερε την Ιρλανδία ή την Σκοτία. Ε, αναφέραμε την δράση των ε, καταστηματαρχών. Ε, έχουμε λοιπόν παραδείγματα με τα οποία αποδεικνύεται ότι η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών μπορεί να μειώσει τη χρήση των πλαστικών σακουλών κατά 80%. Εκεί ακριβώς όπου λαμβάνονται όμως μέτρα. Με το που θα τροποποιηθεί η σχετική οδηγία για τα απόβλητα εκτελεθεί ισχύ. Τα κρατη θα έχουν πλέον στη διάθεσή του τα εργαλεία για αποτελεσματική δράση και θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Ως πρώτο βήμα θα επιλέξουν μέτρο για να μειώσουν την χρήση των πλαστικών σακουλών και να προσθέσουν προκειμένου ότι η οδηγία αντιμετωπίζει στην πηγή του ένα πρόβλημα με τρόπο προληπτικό. Όσο πιο πολλά προληπτικά μέτρα λάβουμε σήμερα, λιγότερα μέτρα θεραπείας θα χρειαστούμε αύριο. Ιδιαίτερα σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα, όπως πολλά, πολλοί βουλευτές ήδη ανέφεραν. Όπως πολλοί επίσης βουλευτές ανέφεραν, πρόκειται για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο απειλεί επίσης, όχι μόνο βεβαίως, αλλά επίσης και το θαλάσσιο περιβάλλον και την ε, θαλάσσια πανίδα. Είναι λοιπόν παγκόσμιο το πρόβλημα, το οποίο απαιτεί παγκόσμια λύση. Σήμερα μιλάμε μόνο για την κατανάλωση των πλαστικών σακουλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο, πολύ ευρύτερο. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους βουλευτές ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του προβλήματος από κοντά. Η νέα οδηγία επιφορτίζει την Κομισιόν με άλλα καθήκοντα, αναπτύξει μεταξύ άλλων μια μεθοδολογία για τους σχετικούς υπολογισμούς της ετήσιας κατακεφαλήν κατανάλωση των ε, λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Πρέπει να προωθήσουμε την κατανάλωση πραγματικά βιοαποδομήσιμων, λιπασματοποιήσιμων σακουλών και να αξιολογήσουμε και τις επιπτώσεις των, οξο, των οξυγονό διασπόμενων σακουλών στο περιβάλλον. Ας κάνουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν για να πετύχουμε την συμμόρφωση και με τις σχετικές προθεσμίες. Η σημερινή μας προσπάθεια είναι σημαντική κίνηση για τη μείωση της σχετική κατανάλωσης και νομίζω απολάβει δημόσιας υποστήριξη. Με την οδηγία αυτή λοιπόν αποδεικνύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε θέματα τα οποία απασχολούν και τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε πιτροπέ. Και τώρα και πάλι κυρία Άουκεν υπήρχε το λόγο ω εισηγητρία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Βέλα. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη μας νίκη κατά αυτόν στην Επιτροπή που είναι κατά του περιβάλλοντος. Η πρώτη, αλόκη και η τελευταία. Είναι η πρώτη μας, είναι μια ιστορική σημασία σήμερα, αφού καταφέραμε να έχουμε τόσο μεγάλη στήριξη από το σώμα αυτό, από τις χώρες μέλη, προκειμένου να μειώσουμε ουσιαστικά τη χρήση των σακουλών αυτών. Και υπάρχει και ευελιξία όχι τόση όσο αρχικά ήθελε η Επιτροπή, γιατί η ευελιξία δεν οδηγούσε πουθενά στην αρχική πρόταση. Ελπίζω λοιπόν, ελπίζω, είμαι χριστιανή, ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά εδώ βέβαια δεν είμαστε μόνο για να ελπίζουμε, αλλά για να κάνουμε. Και κάνουμε πιστεύω με αυτή την οδηγία. Και χαίρομαι που εσείς μας υποσχεθήκατε ότι θα φροντίσετε να εφαρμοστούν όλα όσα αναφέρονται στην οδηγία και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Από τη Δανία έχουμε. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξη. Πριν από δύο μέρες απέφυγα πέντε τέτοιες πλαστικές σακούλες που μου προσφέρθηκαν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό κατά το χρόνο. Καλά στοιχεία λοιπόν, ευελιξία και ας επαναλάβω ότι εδώ δεν μιλάμε για απαγόρευση. Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μιλάμε για μείωση. Και αν τις χρεώσουμε όχι φόρο, χρέωση της κάθε σακούλας. Τότε οι πολίτες, οι καταναλωτές θα το καταλάβουν, θα σκεφτούν «Μα πρέπει να τα πληρώσω αυτά τα ευρώ για να έχω σακούλα». Μήπως να θυμηθώ ότι έχω τσέπες, ότι έχω δικές μου τσάντες, ότι μπορώ να ξεχρησιμοποιήσω τις παλιές μου πλαστικές σακούλες, οπότε να μην πάρω καινούρια. Είναι καλό, είναι θετικό να αλλάξουν συνήθειες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας. Είναι μια ιστορική μέρα η σημερινή και ας μην είναι η τελευταία μας νίκη για το περιβάλλον, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια και εγώ θέλω να συγχαρώ επίσης όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτή την επιτυχία. Έκλεισε λοιπόν η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει σε λιγότερο από μία ώρα από τις 12.30 και μετά. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα.